Έχουμε τη συζήτηση της κυρίας Χιούμπνερ και του κυρίου Λάινεν για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συστήσω σε όλους τους νέους βουλευτές να τηρούν, που τώρα ήρθαν, να τηρούν το χρόνο αγόρευσης, διότι έχουμε καθυστέρηση. Η κυρία Χούμπνερ, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Βρισκόμαστε εδώ διότι αποφασίσαμε να τροποποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Εκλογική Νομοθεσία που ισχύει από το 1976. Εν μεταξύ, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ευρώπη έχει ε, περάσει μεγάλες ε, αφάνταστες αλλαγές τόσο όσον αφορά το πεδίο, το, το, τη δράση της όσο και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έχουμε αλλάξει σε μέγεθος αλλά και όσον αφορά τις αρμοδιότητες ε, αλλά και τον αντίκτυπο των αποφάσεων της Ένωσης ε, στον καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Και άρα λοιπόν δεν είναι εντυπωσιακό το ότι θέλουμε να αλλάξουμε και να προσαρμόσουμε την εκλογική νομοθεσία του 76 στη νέα πραγματικότητα. Και αυτή η έκθεση τονίζει την ε, βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποφασίζει για τη δική του εκλογική διαδικασία. Έχουμε παρόμοιε εμπειρίε ω ευρωβουλευτέ από ευρωεκλογέ που εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά εθνικέ σε περιεχόμενο. Δεν συζητώνται ευρωπαϊκά ζητήματα στη διάρκεια των εκλογικών ε, εκστρατιών. Δεν υπάρχει ορατότητα τη ευρωπαϊκή διάσταση σε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία και γι' αυτό και προτείνουμε να αλλάξει ο εκλογικό νόμο του 1976 στην πρόταση αυτή δίνουμε το δικαίωμα στο Ευρωκοινοβούλιο να αποφασίζει για τη ημερομηνία των εκλογών. Ζητούμε από τα κρατημέλη να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι πολίτε που εργάζονται ή ζουν εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να ψηφίσουν. Επίσης προτείνουμε έναν μηχανισμό για να αποφεύγεται η διπλή ψήφο. Συζητάμε από τα κρατημέλη να δημιουργήσουν τις προδιαγραφές για εκλογές με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του ίντερνετ, μέσω του ταχυδρομείου. Ε, οι άνθρωποι με μειωμένη κινητικότητα σίγουρα θα ωφεληθούν από αυτό και ξέρω ότι ορισμένοι συνάδελφοι ανησυχούν για την ψηφοφορία μέσω ίντερνετ, αλλά μπορεί να γίνει με ασφαλή τρόπο. Έχουμε το παράδειγμα της Εστονίας που άρχισε τις ψηφοφορίες μέσω του ίντερνετ του 2005 όπου το 2% των Εστονών αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο φέτος 30% των Εστονών ψήφισαν μέσω του ίντερνετ Επίση, θέλουμε να έχουμε περισσότερη ισότητα των φύλων στα ψηφοδέλτια. Προτείνουμε διάφορε ευθυγραμμίσει ε, προσθεσμιών για διάφορε εκλογικέ δραστηριότητε, όπω η ε, σύσταση των ψηφοδελτίων. Τα εθνικά κόμματα θα πρέπει να ενημερώνουν τους ψηφοφόρου μέσω των ψηφοδελτίων του την το, το Ευρωπαϊκό Κόμμα στο οποίο ανήκουν. Οι πολίτες θα πρέπει αυτό να γνωρίσουν. Με διάφορες τέτοιες δράσεις ελπίζουμε πως θα συμβάλλουμε ώστε οι ευρωεκλογέ να είναι πραγματικά ευρωπαϊκές και να αυξήσουμε το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη σημαντική φάση της ε, δράσεις στις, ευρω... στις ευρωεκλογές και μέσω της ενήμερης του συμμετοχής στις ευρωεκλογές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάινεν. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μοναδικό παγκόσμια. Πουθενά άλλου δεν έχουν οι πολίτες την δυνατότητα σε 28 κράτη-μέλη μάλιστα να επιλέγουν ένα κοινό κοινοβουλευτικό σώμα που θα τους εκπροσωπεί. Πουθενά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ευρωβουλή. Γνωρίζουμε όμως ότι αυτές οι εκλογές ε, σε 28 κράτη-μέλη πολλά προβλήματα δημιουργούν παρότι οκτώ φορές είχαμε ευρωεκλογές. Δεν έγιναν πολλά πράγματα όμως και υπάρχουν ελλείψεις και κενά σε σχέση με τις ευρωεκλογές που δεν έχουν αρθεί. Γι' αυτό κάνουμε μια νέα προσπάθεια τώρα να υποβάλουμε προτάσεις για τις επόμενες ευρωεκλογές του 2019 δηλαδή ώστε να είναι πιο διαφανείς, πιο δημοκρατικές στο χαρακτήρα, του, στο χαρακτήρα τους και πρέπει να πούμε και πιο ευρωπαϊκές ως εκλογές. Η κυρία συνάδελφος Χιούμπνερ προανέφερε ήδη ότι συστάσεις ε, διατυπώνουμε προς τα κράτη-μέλη και για την εκλογική πράξη του 1976 που θέλουμε να τροποποιηθεί, στι συστάσεις τι λέμε. Θέλουμε η πρόσβαση, η προσπελασιμότητα να διευρυνθεί για τις ευρωεκλογέ. Πιστεύουμε ότι η νέα γενεά πρέπει να προσκληθεί να συμμετάσχει σε αυτέ τι ευρωεκλογέ. Και πολλοί νέοι θα μπορούσαν έτσι για πρώτη φορά με την ηλικία των 16 ετών όταν θα τα ολοκληρώνουν να προσέρχονται στις ευρωεκλογέ. Μια τέτοια συμμετοχή στι εκλογέ θα σφραγίσει μακροπρόθεσμα τι ευρωεκλογέ. Πρέπει να εξετάσουν τα κράτη-μέλη όπω και η Αυστρία να μπορέσουν να μειώσουν την ηλικία των εκλογέων που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχή στις εκλογές στα 16 χρόνια, όπως το έκανε η Αυστρία. Και μπορούμε να προχωρήσουμε σε σχέση, για παράδειγμα, με το να καταλήξουμε στο να προσκαλέσουμε να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές με κάθε τρόπο. Και η επιστολική ψήφος απαγορεύεται σε πολλές χώρες. Δεν είναι όλοι οι πολίτες ε, στο σπίτι τους ε, στις ε, ευρωεκλογές και όλες αυτές οι δράσεις και με την ηλεκτρονική ψήφο μπορούν να βοηθήσουν Είδαμε ότι οι εκλογικοί κατάλογοι λίγες μέρες, ε, κάποιες 17 μέρες κιόλα πριν από τις ευρωεκλογές ε, ολοκληρώνονται. 17 μέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών. Εμείς λέμε τουλάχιστον 12 εβδομάδες. Τρεις μήνες θα ήταν πιο λογικό να μπορούν να κατατίθενται αυτοί, αυτοί οι κατάλογοι, τα, ε, αυτοί οι εκλογικοί συνδυασμοί. Και για τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα έχουμε εθνικές συζητήσεις που που διεξάγονται πολλές φορές αποκλειστικά και χάνεται η ευρωπαϊκή διάσταση στις ευρωεκλογέ. Πρέπει να είναι όμως ευδιάκριτος ο χαρακτήρας αυτών των εκλογών και στα ψηφοδέλτια να, υπάρχουν, να υπάρχει ο λογότυπος ε, να αναγράφεται για την προβολή των πολιτικών ομάδων και κομμάτων η ονομασία και το λογότυπο στα ψηφοδέλτια. Ως ευρωπαϊκά κόμματα να μπορούν να παρουσιάσουν τους ανώτατους υποψηφίους που έχουν και για το αξίωμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως υποψηφίων, ώστε να καθορίζονται αυτά όπως πρέπει. Μια τεράστια πρόοδος θα ήταν η ισότητα των φύλων. 50-50 ή κατά το μισό να είναι γυναίκες οι υποψήφοι ε, σε σχέση με το άλλο ήμιση που θα είναι άντρες. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό. Ήδη το 2019 μπορεί κανείς λένε ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνει κάτι τέτοιο. Το αργότερο μέχρι το 2024 έστω να επιτευχθεί και θέλουμε και η ισότητα να επιτευχθεί οπωσδήποτε. Έχουν ελάχιστα κατόφλια 26 κράτη-μέλη, το 3% για την εκπροσώψη. Γιατί να μην το κάνουν και τα άλλα δύο κράτη-μέλη που απομένουν. Εμείς λέμε λοιπόν 3%. Άλλοι ήθελαν να πάνε πιο πέρα, να έχουμε και πανεθνικούς ε, ε, καταλόγους στα ψηφοδέλτια. Αποφασίσαμε αυτό όμως να κατοχυρωθεί συνενετικά μια και απέτυχε πολλές φορές προηγούμενα το Ευρωκοινοβούλιο και χρειάζεται μια εναλλακτική προσέγγιση και συζήτηση. Ελπίζω ότι θα υπερψηφίσετε λοιπόν συνάδελφοι αυτές τις πραγματιστικές ρεαλιστικές προτάσεις. Κύριε Καρίκε, κατάλαβα σωστά ότι ζητάτε παραπάνω από το χρόνο αγόρευση να μιλήσετε, να θέσετε ερώτηση στα πλαίσια τη γαλάζια Κάρτα, ε, να θέσετε ερώτηση προ τον κύριο Λάινεν. Ναι, ο κύριο Λάινεν δέχεται τη γαλάζια κάρτα. Ορίστε, σα ακούμε. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο αυτό που γίνεται. Κύριε Λάινεν, γνωρίζετε αυτές τις δύο αναλύσεις, αμφότερες και για το Ευρωπαϊκό Εκλογικό Δίκαιο. Μπορείτε ίσως, αν μπορείτε να δείτε ε, ε περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για επαΐοντες ε, για το εκλογικό δίκαιο. Έχουμε μία με ένα σαφές όχι και μία με ένα ναι μία υπέρ, μία κατά. Δεν βρίσκεται ότι είναι αξιοπρόσεκτο να έχουμε δύο πανάκριβες τέτοιες μελέτες με δύο αντιφατικά αντίθετα αποτελέσματα από πλευράς τους. Τι λέτε γι' αυτό, ο κύριος Λάινεν. Κύριε Λάινεν, παρακαλώ. Ναι, αγαπητέ συνάδελφε, έχουμε διαβουλευτεί επ' αυτού επανειλημμένα θεωρούμε ότι η ισότητα των ευκαιριών στην εκλογική διαδικασία πρέπει να διασφαλίζεται στα 28 κράτη-μέλη. Έχουμε σήμερα την κατάσταση σε μία ή δύο χώρες με 0,6% των ψήφων μπορεί κανείς να επιτύχει την διασφάλιση μιας έδρας, ενώ σε άλλες χώρες απαιτείται 3% τουλάχιστον. Αυτό δεν είναι ισόρροπο και αναλογικό. Εμείς είπαμε λοιπόν, αυτή είναι η καινούρια τελευταία δική μας γραμμή και η πλειοψηφία το σχετικά. Κυρία Κρέτσου, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συγγητές, ε, κύριε Λάινεν, κυρία Κούνερ, είναι ιδρυτική αξία η δημοκρατία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασκούν την εξουσία σύμφωνα στι τι προδιαγραφέ τη αντιπροσωπευτικότητα και τη λογοδοσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο μοιράζονται κοινό στόχο. Θέλουν να ενισχύσουν τη δημοκρατική νομιμότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχαίρω το Κοινοβούλιο για την πρόταση τροποποίηση των κανόνων, για την εκλογή των μελών. Ε, κάτι που συζητάτε σήμερα. Η έκθεση που ψηφίστηκε στην Επιτροπή ΑΦΚΟ βάσει της προτάσεως της κυρίας Ντανούτα Χούμπνερ και του κυρίου Ζολάινεν έχει τη δυνατότητα να γίνει ακρογωνίως λίθος στην προσπάθεια ε, αλλαγής του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Ε, είναι κάτι που το αναγνωρίζουμε όλοι, ότι ε, ήταν μια διαδικασία οδυνηρή, πολύ μεγάλο εγχείρημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήξερε ότι έχει ενισχυμένο ρόλο το Ευρωκοινοβούλιο όσον αφορά το διορισμό του Πρόεδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τι συνθήκε τη και άκουσε και τι εκκλήσει του Κοινοβουλίου και ζήτησε τα πολιτικά κόμματα να καθορίσουν στελέχη για, τον, για να κρίνουν το διορισμό ε, του Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για πρώτη φορά οι πολιτικές οικογένειες πρότειναν κάποιον και ο κ. Ζαν Κλοντ σαν υποψήφιο συνέλεξε την πλειοψηφία ε, των ψήφων στο Ευρωκοινοβούλιο και διορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εξελέγει από το Ευρωκοινοβούλιο σαν πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι καινοτομία αυτή των εκλογών του 2014. Οπότε η εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεδέθη πιο στενά με τους εκλογείς. Και στις μελλοντικές εκλογές θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το στοιχείο. Έτσι θα αυξηθεί η δημοκρατική νομιμότητα τη διαδικασία λήψη των αποφάσεων στην Ευρώπη. Σημαντικό βήμα πρόοδου για να υπάρχει μια πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική σφαίρα. Προτείναμε μεταρρύθμιση σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσουμε την πολιτική λογοδοσία. Τα ευρωπαϊκά κόμματα θα πρέπει να καθορίσουν του υποψηφίου του τουλάχιστον 12 εβδομάδες των εκλογών. Οι μεταρρυθμίσει μπορεί να βοηθήσουν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ πολιτικών διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο και θα δείξουν τη σχέση μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στα ψηφοδέλτια και στις πολιτικές εκπομπές την προκλητική περίοδο. Έτσι θα υπήρχε σχετισμός μεταξύ των διαφόρων φορέων και θα βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων στη διαδικασία. Όλοι υπήρξαμε θύματα της έλλειψης συζητήσεων για τα ευρωπαϊκά θέματα. Και είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό τα εθνικά πολιτικά κόμματα και οι εθνικές αρχές έχουν αποφασιστικό ρόλο να παίξουν. Θα μπορέσουν να βελτιώσουν τη διαφάνεια, να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες, να γνωρίσουν τις ε, ευρωπαϊκές συνέπειες που έχουν οι ψηφοφορείς σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να διοργανώνονται οι ευρωπαϊκές εκλογές βάσει προδιαγραφών. Ελάχιστο όριο σε κράτη-μέλη για τον επιμερισμό των εδρών. Έτσι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε και την ευρωπαϊκή διάσταση των εκλογών πρέπει να έχουμε ένα ελάχιστο κατόφλιο. Έτσι το Ευρωκοινοβούλιο θα είναι αποτελεσματικότερο. Θα μειωθεί ο κίνδυνος κατακαιρματισμού και θα διευρυνθούν οι, θα, οι σταθερές πλειοψηφίες. Μιλάμε για την κρίση της αντιπροσωπτικής δημοκρατίας για την απογοήτευση των ανθρώπων εναντί της πολιτικής. Το να προωθήσουμε τη συμμετοχή είναι σημαντικό για να προωθηθεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Γι' αυτό καλωσορίζω ένθερμα τις προτάσεις για επέκταση ε, τη ψηφοφορία για υπηκόου τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ζουν σε τρίτε χώρε. Θέλουμε πιο ευέλικτη προσέγγιση για την ε, ψηφοφορία. Για να προωθήσουμε την συμμετοχή τη μεγαλύτερη των γυναικών στις ευρωεκλογέ με εκλογικού καταλόγους που πετυχαίνουν την ισότητα των φύλων. Κάτι που προτείνεται στην έκθεση. Είναι σημαντικό βήμα αυτό στη σωστή κατεύθυνση. Ήμουν εδώ, αλλά στην άλλη πλευρά, στην άλλη όχθη, όταν είχα προτείνει υποσωστώσεις. και πρέπει να κάνουμε κάτι σε εθνικό επίπεδο, γνωρίζοντα τα τη χώρα μου τα λέω αυτά. Σε πολλέ χώρε είναι καταστροφική κατάσταση σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση και σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων. Τουλάχιστον εδώ εφαρμόζουμε αυτή την αρχή που είναι πολύ σημαντική. Θέλουμε δίκαιη και αντικειμενική κάλυψη από τα ΜΜΕ στην προεκλογική περίοδο. Βασικό στοιχείο αυτό. Το τονίζω αυτό είναι σημαντική προϋπόθεση για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Σημειώνω την πρότασή σας να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή εκλογική αρχή. Σε κεντρικό επίπεδο να τίθεται πληροφορίε για τι ευρωεκλογέ. Θα πρέπει αυτό, πριν αναλυθούν υποχρεώσει, να εξεταστεί προσεκτικά. Πρέπει να εξετάσουμε τη σκοπιμότητα μια τέτοια προτάσεω. Και ποιε θα είναι οι ευθύνε μια τέτοια αρχή. Ποιε διευθετήσει απαιτούνται για να δημιουργηθεί. θέματα θεσμικά, νομικά, οικονομικά, τι απαιτούνται για να λειτουργήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου να υιοθετηθεί αυτό έγκαιρα. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε τις ομιλίες εκ μέρους των ομάδων. Ο κ. Σέφλιν για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Δεν ε, υπάρχει τίποτα το παράξενο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να θεσπίσει ένα κοινό ελεκλογικό σύστημα για τον εαυτό του. Κάθε, κάθε κοινοβούλιο στον κόσμο το κάνει αυτό. Ένα σύστημα μέσω του οποίου οι πολίτες επιλέγουν τους εκπροσώπους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, παρόμοιο στις χώρες, ε, αν και ε, όχι απόλυτα ίδιο. Το λεπτό ζήτημα εδώ είναι το θέμα του κατοφλίου. Αν θα έπρεπε να υπάρχει δηλαδή ένα ελάχιστο όριο ψήφων που θα πρέπει κανείς να φτάσει πριν να μπορεί να εκπροσωπήσει τους πολίτες. Σε κάποια κατεμέλη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά εν γέννη είναι αποδεκτή πολιτική και πρακτική. Αυτό το κατόφλι έχει στόχο να κρατήσει εκτός ε, τους ε, όχι πολύ σοβαρούς ε, υποψηφίους. Από την άλλη πλευρά μπορεί να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά ψηλό όριο για την είσοδο κάποιου. Ε, ένα κατόφλι αλλά όχι πολύ ψηλό. Αυτό θα ήταν η καλή ισορροπία και αυτό προσπαθεί να φτιάξει αυτή η έκθεση. Να θεσπιστεί ένα κατόφλι αλλά όχι εξεπέραστο. Από κάθε άποψη αυτό, ε, αυτή είναι μια λογική λύση. Σας ευχαριστώ η κυρία Μπρέσο, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών για μέση λεπτό. Σας ευχαριστώ. Ε, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές για το ε, έργο τους, είναι περίπλοκο, ε, και την Επίτροπο για την υποστήριξη που προσέφερε στη δική μας πρωτοβουλία. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό, γιατί είναι μια από τις δύο εκείνες της περιπτώσεις όπου το Κοινοβούλιο έχει νομοθετική πρωτοβουλία, έχει δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας. Εμείς προτείνουμε κάποιες περιορισμένες αλλαγές στην νομοθεσία. Θα ήθελα να θυμίσω ότι από το 1976 το Συμβούλιο αρνείται να αλλάξει το κείμενο του εκλογικού νόμου και άρα να καταστήσει πιο ευρωπαϊκές τις εκλογές, όπως ήδη θύμισε ο συνάδελφος Σέφλινγκ. Οι προτάσεις ε, λοιπόν είναι προτάσεις ε, που είναι περιορισμένες αλλά που στόχο έχουν το να έχουμε μια πιο ομοιογενή ε, εκλογική νομοθεσία. Να σας θυμίσω κάποιες προτάσεις όπως αυτή που στόχο έχει να δώσει η ορατότητα στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και άρα να δώσει και ευρωπαϊκό νόημα στις εκλογές, να σταθεροποιήσει τον ορισμό των υποψηφίων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να επιτρέψει να τους γνωρίζουν οι εκλογείς μέσω ενός κατάλληλου αριθμού εβδομάδων, στη διάρκεια των οποίων θα είναι γνωστά τα ονόματα, έπειτα εξισορρόπηση των φύλων που πιστεύω είναι απαραίτητη, ε, το θέμα των διακρατικών ψηφοδελτίων που θα μπορούσε να ξανατοποθετηθεί, τουλάχιστον με ένα εκτιμώντα, δηλαδή ε, μια μικρή σημείωση. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε για πρώτη φορά μια, έναν εκλογικό νόμο εδώ, στο, το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριο Ουιαντόφσκι για δύο λεπτά εξ ονόματος της CCR. Κυρία Πρόεδρε, ε, η CR ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί το εκλογικό δίκαιο για τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ε, θετικό. Δεν βλέπουμε να υπάρχει ανάγκη κάποιων τροποποιήσεων, ιδιαίτερα κάποιων τροποποιήσεων για το, την ενοποίηση και κεντρική διαμόρφωση του εκλογικού δικαίου. Δύο πράγματα όμως πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτον, όταν πρόκειται για την ηλικία που θέλουμε, προτείνεται να μειωθεί στα 16 έτη για τους εκλογείς ή αν προτιθέμεθα να ε, δεχθούμε εκλογή ε, από τους πολίτες μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου, του διαδικτύου. Δεν είμαστε πεισμένοι για αυτά. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση η εκλογική διαδικασία και δεν είναι το ίδιο όπως ένα βήμα ηλεκτρονικής έκφρασης ε, όπως το διαδίκτυο. Ακόμα πιο σοβαρή είναι η σκέψη μιας ε, ενοποίησης και ενιαίας διαμόρφωσης υποκεντρικής πρακτικό χαρακτήρα σχεδιασμού του εκλογικού δικαίου να υπάρχει για παράδειγμα να υπάρχουν υποχρεωτικά ε, στοιχεία τα οποία θα είναι υποχρεωτικά όπως ε, το ολογότυπος. δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν τέτοια πράγματα τα πολιτικά κόμματα τα οποία υφίστανται στα κράτη-μέλη μας ε, και τα οποία συμμετέχουν και μπορούν να δρουν θα μπορούν αυτά να υποβάλουν τις προτάσεις τους για να εκλεγούν στο Ευρωπαϊκό, Δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά πρέπει να ισχύουν όμως από κοινού για όλους όλους και με βάση αυτές τις αρχές θα πρέπει να δράσουμε με σεβασμό των συνταγματικών παραδόσεων των κρατών μελών. Όσο περισσότερο βρισκόμαστε πιο κοντά στα κράτη μας, στα έθνη μας και στα όσα ισχύουν εκεί, τόσο πιο αποτελεσματικοί θα είμαστε ένας κεντρικός σχεδιασμός θα σημαίνει ότι όλο και περισσότερο θα αποκλίνει και θα απομακρύνεται το Ευρωκοινοβούλιο από τους πολίτες. Γι' αυτό θα καταψηφίσουμε αυτή την έκθεση. Ορτώντα Παγάς, Ορτώντα Ρουίς. Μάλιστα πρόεδρε σας ευχαριστώ. Σε αυτή τη συζήτηση αποφασίστηκε να καθυστερήσει η ψηφοφορία ώστε να υπάρξει χρόνος να αναλυθούν κάποιες από τις πτυχές που συναπαρτίζουν την έκθεση και που θα μπορούσαν ίσως να την συμπληρώνουμε. Ήταν λίγο φιλόδοξη η διαδικασία μεταρρύθμισης μέχρι σήμερα. Είναι ανεπαρκής ίσως χρήση δυνατοτήτων ή υπερβολικά συνετή δραστηριοποίηση και βρισκόμαστε σε μια κρίση που υπονομεύει τις, ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Μόνο ένα ε, σε, κάθε τέσσερις ε, συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές και βλέπουμε και το τι συμβαίνει στις ε, εθνικές εκλογές που καθορίζουν διότι οι κυβερνήσεις τα μεγάλα κόμματα έτσι ε, ε, δρούν. Υπάρχει όμως διχασμός μεταξύ εκείνων που λέγουν στο Ευρωκοινοβούλιο και ιδιαίτερα εκείνων που πράττουν στις χώρες τους τα κόμματα αυτά όταν κυβερνούν θα πρέπει πραγματικά να δούμε τι μπορεί να γίνει με την συνειδητοποίηση από πλευράς ε, ευρωπαϊκών εκλογών. Οι ευρωπαϊκές εκλογές θα μπορούσαν να είναι κάτι παραπάνω από την αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών και μπορούν να προσεγγίσουν το όργανο, το θεσμικό αυτό όργανο στους πολίτες. Και οι εκπρόσωποι θα πρέπει να υποβαλόμεθα στην λογοδοσία διαρκώς. Πρέπει να διαρωτηθούμε αν αυτή η έκθεση επιτυγχάνει πραγματικά αυτούς τους στόχους με τις συστάσεις της. Ε. Εμείς πιστεύουμε περισσότερο ότι υπάρχουν μεν αλλαγές που είναι θετικές, κάποιες άλλες που είναι εξοραϊστικές ε, αλλαγές ε, και κάποιες άλλες που δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν. Έχει βελτιώσει η έκθεση όσον αφορά την ισότητα του φύλου ή την ψήφιση τη συμμετοχή στις ευρωεκλογέ από πολίτες που ζουν σε τρίτα κράτη. Όμως δεν μπορεί να υπάρξει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά για παράδειγμα τα ψηφοδέλτια. Εκεί υπάρχουν ελλείψεις. Οι τροποποιήσεις είναι ίσονος σημασία. και θεωρούμε ότι δεν ενισχύεται έτσι μια μεγαλύτερη δυνατότητα ενοποίησης και ολοκλήρωσης όπως απαιτείται. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σόλτ, παρακαλώ, εξ ονόματος της Ενωτικής Αριστεράς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πίτροπε, μετά τις εκλογές, πριν από τις εκλογές αγαπητοί συνάδελφοι και υπεραιτέρω περαιτέρω μεταξέλιξη του Ευρωπαϊκού Εκλογικού Δικαίου βρίσκεται και έχει ενταχθεί σωστά πιστεύουμε στην δική μας ημερήσια διάταξη εργασιών. Πολλά μπορεί να επιτύχει, όμως πρέπει να μετρηθεί με γνώμονα εκείνων που θα επιτελέσει μπορεί να υλοποιήσει αυτά τα οποία απαιτούνται σε σχέση με την απομάκρυση των πολιτών από την πολιτική. Μπορεί να δώσει δυνατότητες ενεργού συμμετοχή σε σχέση με την παθητική αντιμετώπιση μέχρι σήμερα. Η μεγάλη έλλειψη αυτής της έκθεσης, αγαπητέ εισηγητά και συνεισηγήτρια, με όλες τις καλές προθέσεις πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι έγκυται κυρίως στο ότι δεν είναι ιδιαίτερα θαραλέα η προσέγγιση για τις μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που απαιτούνται σε σχέση δηλαδή με το Συμβούλιο. Δεν ακολουθεί λοιπόν τις φιλοδοξίες ε, για περισσότερο ευρύτερο ρόλο και μεγαλύτερες δυνατότητες. Προσπαθεί περισσότερο τεχνικές δυνατότητες να χειριστεί που δεν είναι αποτελεσματικές. Η ειδική δυναμική της ίδιας, της κοινωνίας και των πολιτών πρέπει να αποτελέσει θεμέλιο. Οι ε, δημοκρατικές αλλαγές δεν μπορούν να γραμμίζονται με αυτές τις προτάσεις σε σχέση με τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρώπης. Για παράδειγμα με τη μεγάλη συμπολίτευση στη Γερμανία. Αναφέρθηκε ότι εδώ πραγματικά μπορεί να αποτελέσει αυτό ίσως πρόκληση για την κατάσταση πραγμάτων που υφίσταται σήμερα. Ευχαριστώ. Euh, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η μεταρρύθμιση του εκλογικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το γεγονός ότι είχαμε δύο εισηγητές για αυτή την έκθεση είναι ένα πρώτο μήνυμα για την ε, ε, σύμπραξη όσον αφορά τις ε, προτάσεις που υποβάλλονται. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει και κάποια έλλειψη ελαστικότητας όταν η συζήτηση κατέληξε στο να γίνουν δεκτές ή όχι κάποιες από τις προτάσεις και συστάσεις που υπευλήθησαν από άλλες ομάδες. Γι' αυτό λυπούμε πολύ να πω ότι είναι μια αποδυναμωμένη έκθεση που δεν ήταν σε θέση να μπορέσει να αρθεί στο ύψος των ιστορικών προκλήσεων. Μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων θα έπρεπε να ενδυναμώνει την ουσία της συμμετοχής ε, των ε, πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν τα κατάφερε όμως. Και πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής τέσσερις ε, τομείς ένα υποχρεωτικό κατόφλι που είναι σαφώς απαράδεκτο σε σχέση με τον γερμανικό συνταγματικό κώδικα και τώρα θα θεωρείται υποχρεωτικό για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πραγματικά αντιβαίνει στην προστασία των μειονοτήτων. Δύο, ε, διεθνική υπερεθνικά ε, ψηφοδέλτια. Ήδη αυτό ε, σε, ένα απλό, σε μια απλή αιτιολογική σκέψη αντανακλάται. Η εισαγωγή της ισότητας των Αναβλήθηκε και αυτό μέχρι τις ευρωεκλογές του 2024. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μέχρι τότε. Θέσπιση ελάχιστη ηλικία στα 16 έτη. Εκεί παραμείναμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε James, του Άκουσα τις δηλώσεις που περιέγραφαν τους προτινόμενους στόχους και έγινε προσπάθεια να δικαιολογηθούν. Ειλικρινά, με έκπληξη άκουσα αυτά που άκουσα. Υπάρχει ο Τζορτζ Όρουελ, φημισμένο συγγραφέα. Θα ήταν υπερήφανο αυτών που περιγράφησαν, για αυτά περιγράφησαν απόψε. Και για εκείνου που είχαν τρομοκρατηθεί από το βιβλίο θα είχαν βρει βάση για του φόβου του εδώ αυτά που άκουσαν. Λοιπόν, λιγότερη δημοκρατία παρά εκκλήσει για κάτι τέτοιο και περισσότερα εκλογικά αποτελέσματα ήταν ο στόχο. Κοιτάξτε τι έγινε στην Πορτογαλία πρόσφατα όσον αφορά τι εκλογέ και τα αποτελέσματα των εκλογών. Στόχο ποιο είναι. Περισσότερα από αυτά που άκουσα απόψε και περισσότερα από αυτά που περιγράφησαν, δηλαδή να αγνοείται η βούληση του λαού, να αγνοείται το δημοκρατικό αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν άκουσα μέχρι τώρα καμία περιγραφή τη κλίμακα των παγκοσμίων ε, επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και τη κλοπή ταυτότητα. Και έχουμε εστιαστεί στι προσπάθειε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα κλείσω λέγοντα ότι ο εκλογικό νόμο είναι θέμα που αφορά κυρίαρχα κράτη και όχι αυτό το κοινοβούλιο. Είναι ξένο για αυτά τα θέματα το Ευρωκοινοβούλιο. Ο κύριο Άνεμαν για ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, ο εκλογικό νόμος που χρονολογείται από το 1977 αρκεί για τη διεξαγωγή εκλογών στα κράτη-μέλη του 1976. Θέλουμε να ε, ε, εκλέξουμε τώρα έναν καινούριο εκλογικό νόμο, ώστε το εκλογικό σώμα το ευρωπαϊκό να ψηφίζει μαζικά και θα υπορροφηθούν οι ψηφοφόροι να υποστηρίξουν τη νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ θα παραγωνίζονται τα κράτη-μέλη. Ε, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αφαιρεί πολλά δικαιώματα των κρατών μελών. Οι βουλευτέ δεν θα εκπροσωπούν πλέον τι χώρε του, αλλά όλου του πολίτε Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ταυτόχρονα θα, υπάρχει, θα εισαχθεί υποχρεωτική ψηφοφορία παντού, ώστε να αποφευθεί περαιτέρω κατακαιρματισμό του εκλογικού σώματος και θα μπορούν να ψηφίζουν οι λαοί και για μικρά κυρίως αντιευρωπαϊκά ε, κόμματα. Θέλουμε κάθε χώρα να μπορεί να αποφασίσει από μόνη της ε, τι διαδικασία θέλει να ακολουθήσει για του πολίτε τη. Έχετε μια γαλάζια κάρτα. Εγώ θα σας κατακεραυνώσω. Θα είμαι πάρα πολύ γρήγορα μάλλον. Λοιπόν, ε, εμείς εκπροσωπούμε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τις χώρες μας εδώ. Θα ήθελα να ξέρω αν έχετε επίγνωση αυτού. Τι εκπροσωπούμε δηλαδή εμείς εδώ. Απάντηση. Κυρία Βουλευτά, Όσον αφορά το περιεχόμενο των ε, συνθήκων, δεν εκλέγομαι γι' αυτό. Βλέπετε τι σημαίε που έχω γύρω μου και θα βλέπετε να φυτρώνω όλο και περισσότερε σημαίε. Εκπροσωπούμε τι εκλογέ που μα ε, ψήφισαν. Έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Και εσεί έχετε δικαίωμα να υποκρίνεστε ότι εκπροσωπείτε όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν ισχύει όμω. Εμεί εκπροσωπούμε του δικού μα ψηφοφόρου, του λαού μα και τελικά την Ευρώπη. Ο κύριο Βόμποντα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε η σύμβαση για την συνθήκη για λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την δυνατότητα της τροποποίησης του εκλογικού δικαίου και ανάληψης πρωτοβουλίας για αυτή την αλλαγή. Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι επετεύχθη σε σχέση με την Επιτροπή Συνταγματοθέσεων να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυνατότητα και να δράσουμε όπως έπρεπε. Η ιδέα η οποία ενέπνευσε την έκθεση πρέπει να υποστηριχθεί η ενδυνάμωση με άλλα λόγια των ε, δημοκρατικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η αφετηρία για την θετική αντιμετώπιση των ευρωεκλογών και αυτό ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε μια υψηλότερη συμμετοχή των πολιτών στις ευρωεκλογές και αυτό θα έχει θετική έκβαση συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δημοκρατικό δημιούργημα το Ευρωκοινοβούλιο και πρέπει να ανταποκρίνεται στην ανάγκη να διευρύνεται και να προάγεται το ευρωπαϊκό πνεύμα είναι προς το συμφέρον μας λοιπόν να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας και να μπορέσουμε να τηρήσουμε τα υπεσχημένα και γι' αυτό υποστηρίζω αυτή την προσέγγιση. Ο κ. Σίλβε Περέιρα για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κανονικά αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο στο να ε, θρυνούμε για το παλιό πρόβλημα του δημοκρατικού ελλείμματος ε, από ότι στο να συζητούμε μέτρα για να βελτιώσουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες μας. Γι' αυτό και θέλω να χαιρετήσω τους δύο συναδέλφους, Λάινεν και Χούμπνερ, για την εξαιρετική τους έκθεση που προτείνει μια, έκθεση που προτείνει μια πολύ καλή και ρεαλιστική μεταρρύθμιση για τους ευρωπαϊκούς, την Ευρωπαϊκή Εκλογική Νομοθεσία. Είναι από τους λίγους νομίζω όπου το Ευρωκοινοβούλιο έχει δικαίωμα για νομοθετική πρωτοβουλία. Έχουμε το καθήκον ε, και όχι μόνο το δικαίωμα να βελτιώσουμε τα πράγματα. Ήδη κάναμε ένα σημαντικό βήμα στο να τις ευρωεκλογέ με τι υποψηφιότητε του Προέδρου τη Κομισιόν και πρέπει τώρα να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο με αυτή τη μεταρρύθμιση τα υλικά της εκστρατείας και τα ψηφοδέλτια θα, δίνουν περισσότερο ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Θα έχουμε τις ίδιες προθεσμίες για την υποβολή των ψηφοδελτίων και των υποψηφίων. Τις ίδια ωράρια για να ψηφίσουμε την ίδια δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου και έχουμε και μια ρήτρα ε, που απαιτεί 3 με 25.000 ε, ψήφους για να εκλεγούν οι υποψήφοι κρατών που έχουν πάνω από 25 βουλευτές. Σαφήνεια έτσι ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ποιον ψηφίζουν και για ποιο λόγο. Έτσι η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία θα είναι καλύτερη αν γίνει αυτή η εκλογική μεταρρύθμιση. Κυρία Πρόεδρε, το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο το 5% ε, κατόφλι το θεώρησε αντισυνταγματικό για συμμετοχή μικρών κομμάτων στο σώμα και φυσικά ε, αυτό ε, οδήγησε στο ότι η S5 η Χριστιανοκοινωνική Ένωση και οι πράσινοι θέλουν ε, να τροποποιήσουν τα πράγματα ώστε να ενισχυθούν λέει με τα μικρότερα κόμματα όμως αυτή η προσέγγιση απερίφθη και το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο ανέφερε σε σχέση με τον κύριο Λάμστορφ για παράδειγμα της FDP ότι αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να γίνουν να είμαστε ειλικρινεί. Ε, τα θνησιγενή επιχειρήματα μόνο ανταλλάξατε με αυτόν τον τρόπο και θέλατε να παρακολύσετε αυτή τη δυνατότητα ώστε να υπάρχει ένας τέτοιος φραγμός ε, για το εκλογικό δίκαιο και να αποκλειστεί το συνταγματικό ε, το... η συνταγματική εκπροσώπηση των μικρών κομμάτων. Αυτό είναι βλαπτικό κύριε Λάινεν. Κυρία Μίλλερ για ένα λεπτό. Με μεγάλη πλειοψηφία εδώ λοιπόν στο Ευρωκοινοβούλιο η τροποποίηση, η μεγάλη μεταρρύθμιση του εκλογικού δικαίου λέει θα επιτευχθεί. Και ενώ πάντα βρισκόταν η αρχή της επικουρικότητας στο επίκεντρο, για μένα δεν υπάρχει κανένας λόγο να εισαχθεί ένα κατόφλι 3% διότι μόνο σε δύο από τα κράτη-μέλη στην Ισπανία και τη Γερμανία ε, βλέπουμε κάτι τέτοιο θα είχε επίπτωση. Και το επιχείρημα αυτό για τις μικρές ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει και μπορούν εύκολα να υπάρξουν αντεπιχειρήματα. Έχουμε αποφάσεις ε, του συνταγματικού δικαστηρίου κατά του κατοφλίου αυτού και εδώ θέλετε να παρακάμψετε αυτές τις ε, αποφάσεις. Αυτό θα οδηγούσε αν συνέβαινε, αν ενεκρίνεται 8 εκατομμύρια ψήφοι να μην μπορούν να έχουν εκπροσώπηση κοινοβουλευτική. Εγώ μπορώ να πω ότι οι ευρωβουλευτές εδώ με, τους, με τις περισσότερες ψήφους είμαι εγώ εκείνη και έχω 1,6% στη χώρα μου περισσότεροι δηλαδή πολίτες από ότι οι κάτοικοι της Μάλτας ε, με υπεψήφισαν έχω κάθε νομιμότητα λοιπόν να λέω αυτά που ανέφερα ο κ. για ένα λεπτό. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο κυρία Πρόεδρε. Η εισαγωγή ενός κατοφλίου 3%, 3% ή 5% αφορά μόνο τη Γερμανία και την Ισπανία όπως προαναφέρθηκε διότι είναι οι μόνες χώρες που αφενός έχουν πάνω από 26 ε, ευρωβουλευτές ε, και δεν, δεν υπάρχει ε, μια τέτοια δυνατότητα αποκλεισμού. Τι θα σήμαινε αν υπήρχε μια τέτοια δυνατότητα. Έναντι της δικαιοσύνης για τις μικρότερες ομάδες δεν θα μπορούσε να γίνει λόγος. Ας δούμε τα, τους αριθμούς. 3% στο Λουξεμβούργο είναι 12 περίπου χιλιάδες εκλογείς. 3% στη Γερμανία είναι το 10 πλάσιο αυτών των 12 12.000 του Λουξεμβούργου. Αν πάρει κανείς τους βουλευτέ σε σχέση με αυτή την αναλογία, τότε θα ήταν τριακονταπλάσια η διαφορά. Δημοκρατία το αποκαλείται αυτό. Και οι ψήφοι των μικρότερων κομμάτων θα εντασσόντουσαν στι μεγαλύτερε στα μεγαλύτερα κόμματα που θα υποφελούνται. Αυτά θέλουν να κερδίσουν ψήφου από τα μικρότερα κόμματα. Κυρία Μάιερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα αντιμετωπίζουμε μία από τις πολλές προσπάθειες του Ευρωκοινοβουλίου να λύσει αυτό το θέμα. Υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα των Βρυξελών, παίρνει εξουσία από τα κράτη-μέλη. Βλέπετε τι γίνεται με τη συμμετοχή σε εκλογές. Κανείς δεν ξέρει από τον κόσμο ποιος είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα. Δεν μπορεί να λυθεί αυτό με την απαγόρευση των δημοσκοπήσεων στα κράτη-μέλη, με τη μείωση της δημοκρατίας στα κράτη-μέλη, με το να, να καθορίζουμε όρια κλπ. Ε, γιατί δεν νοιάζεται κανείς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό πρέπει να διορθωθούμε. Γιατί 42% μόνο 42% του λαού ψηφίζει στις ευρωεκλογέ. Η πλειοψηφία των εκπροσώπων των λαών ε, στο Ευρωκοινοβούλιο υποστηρίζουν τις αντιδημοκρατικές απόπειρες. Κυρία Πρόεδρε, οι εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο είναι εκλογές για εθνικούς εκπροσώπους. Στην περίπτωση μου πιστεύω ότι πρέπει να εκπροσωπούμε το λαό της Ολλανδίας. Αυτές οι εκλογές διεξάγονται στην Ολλανδία και τίποτα δεν έχετε. Διακόπτη η κυρία Πρόεδρος, επόμενος ο κύριος Πρέντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θέλω να εκφράσω συγχαρητήρια προς την κυρία Χρύμνερ και τον Γιώ είναι η δεύτερη προσπάθεια μεταρρύθμισης των εκλογικών διαδικασιών και βλέπουμε ότι κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία δεν ήταν καθόλου εύκολο να εξευρεθεί μια ισορροπία μεταξύ φιλοδοξιών και εφικτότητας και πραγματικής εφαρμογής. Τώρα θέλουμε να τα καταφέρουμε η ευρωπαϊκή νομοθετική προσπάθεια δεν είναι μόνο το άθροισμα 28 διαδικασιών κρατών μελών. Γι' αυτό πρέπει οι προτάσεις που εμπεριέχονται στην έκθεση Hübner-Leinen να υποστηριχθούν και πρέπει επιπλέον τις κατευθυντήριες γραμμές ε, να τις τηρήσουμε όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Διότι είναι σημαντικό να υπάρξει περισσότερη Ευρώπη από τις ευρωεκλογέ μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Να αναβαθμιστεί η δημοκρατική νομιμότητα μέσω των εκλογικών διεργασιών. Θέλω να αναφέρω τρία θέματα που είναι σημαντικά για μένα και υπεστήριξα. Η δυνατότητα να ψηφίζουν οι πολίτες από το 16ο έτος της ηλικίας τους. Να υπάρχει δημοκρατική διαδικασία στο διορισμό των υποψηφίων και εισαγωγή ηλεκτρονικής ψήφου και η απλούστευση αυτών των δυνατοτήτων θα δώσει τη δυνατότητα περισσότεροι πολίτες να μπορούν να συμμετέχουν στις ευρωεκλογέ. Ο μεγάλος αριθμός των τροπολογιών ελπίζω ότι δεν θα αλλοιώσει την ισορροπημένη αυτή δομή της έκθεσης. Κύριε Σωτόντο για ένα μισή λεπτό. Μάλιστα κυρίε και κύριοι, η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω. Δεν θεωρείτε ότι 40 χρόνια κυρίε και κύριοι μετά πρέπει να αλλάξει το νομικό ε, πλαίσιο, ο νόμος. Ο νόμος είναι του 1976. Άλλαξε η Ευρώπη αυτά τα 40 χρόνια. Πιστεύω ότι άλλαξε και σημαντικά. Εμείς που είμαστε εδώ παρόντες ε, για τους ίδιους κανόνες πρέπει να έχουμε και τα ίδια δικαιώματα. Θα πρέπει να έχουμε ένα εναρμονισμένο σύστημα εκλογικού δικαίου για τις εκλογές μας, ε, για την εκλογή μας. Δεν θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει εκπροσώπηση των ευρωπαϊκών κομμάτων όχι των εθνικών κομμάτων και των παραρτημάτων τους. Εμείς που, είμαστε, που βρισκόμαστε εδώ εκπροσωπούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών ως Ευρωπαίοι Ευρωβουλευτές. Θα πρέπει να έχουμε κοινούς κανόνες, έτσι δεν είναι, για να βρισκόμαστε εδώ και να δρούμε στο Ευρωκοινοβούλιο με υπερεθνικούς καταλόγους και ψηφοδέλτια, ώστε κάθε κόμμα να έχει την δυνατότητα να έχει εκείνους ως υποψηφίους που θα Πρόκειται να κυβερνήσουν στην Ευρώπη. Δεν είναι λογικό αυτός κανόνας. Και τελευταία ερώτηση προς τους συναδέλφους των Πρασίνων και της Ενωτικής Αριστεράς. Παρακαλώ μην προσθεθείτε εσείς με το όχι στους αντίθετους σε ένα νόμο που δεν είναι τέλειος. Σε ένα νόμο που θα θέλαμε να ήταν καλύτερος. Δεν αξίζει το όχι σας όμως την απόρριψή σας. Αποκινούμε εκείνους που απορρίπτουν την Ευρώπη. Κύριε Ραντουγκί ε, δέχεστε μια γαλάζια κάρτα. Δέχεστε γαλάζια κάρτα από τον κύριο Λεμπρετόν. Ε, 30 δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σα, ορίστε. Σα Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να θέσω αυτή την ερώτηση με την μπλε κάρτα. Με εντυπωσίασε ε, που βλέπετε, που λέτε μάλλον ότι εδώ εμείς δεν αντιπροσωπεύουμε τους ε, λαούς, αλλά θέλετε να αντιπροσωπεύουμε τα ευρωπαϊκά κόμματα. Εγώ προσωπικά πιστεύω πως είναι λάθος αυτό. Η τελευταία ευκαιρία που μας μένει για να λυσώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να τη συμφιλειώσουμε και πάλι με τους λαούς. Εγώ είμαι υπέρ τη διάλυσης τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να τη λύσετε, πιστεύω ότι πρέπει να τη συμβιλίωσετε και πάλι με την Ευρώπη. Εσεί, τι πιστεύετε, δεν είναι αυτή η τελευταία δυνατότητα, η τελευταία ευκαιρία ψασμένη. Ναι, αλλά... Όμως οι λαοί, τα έθνη, είναι η Ευρώπη. Καθώ είναι έθνη αυτοί οι πολίτε είναι Ευρώπη. Θέλω περισσότερα ευρωπαϊκά κόμματα. Δεν θέλω ένα συνονθήλευμα εθνικών κομμάτων. Θέλω ευρωπαϊκά κόμματα που θα εκπροσωπούν τα κυρίαρχα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών πολιτών. Γι' αυτό χρειάζονται περισσότερα ψηφοδέλτια υπερεθνικά και ε, κόμματα ευρωπαϊκά. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, οπωσδήποτε. Γκέρικ, ένα λεπτό. Η S5, η CDU και η CSU είναι κυρίαρχοι στην κατάχρηση της επανεισαγωγής ενός φραγμού 3% και της απόλυτης άγνοιας ε, και παραμέλησης της ε, νομολογίας και της απόφασης του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Δεν έχετε θάρρος. Μία συνάδελφος της CSU λέει παρακολουθούμε τώρα, δηλαδή υπάρχει υπο, εκτίμηση. Ε, όμως οι εκλογείς γνωρίζουν και εκτιμούν. Αυτό είναι η περίπτωση αστερίξ, της αρχής αστερίξ και αυτό γιατί. Διότι περισσότερες εκθέσεις παρακολούθησα εγώ και ε, συνόδεψα από ότι διάφοροι συνάδελφοι κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. Διότι τις, τα μελήματα των πολιτών τα παίρνω σα σοβαρά σε ευρύτερη κλίμακα και με, υψώνω τη φωνή μου για τις οικογένειες. Αν παίρνετε κι εσείς ε, εξίσου σοβαρά τη δουλειά σας όπως ε, και εγώ, πάψτε να κάνετε αυτά τα κόλπα. Πάψτε να αγνοείτε την απόφαση του συνταγματικού γερμανικού δικαστηρίου. Πάψτε να ποδοπατείτε κατάφορα τα δικαιώματα των μικρών κομμάτων και των μικρότερων. Τώρα μπαίνουμε στη φάση του Κατσεδιάη. έχουμε έξι αιτήματα. Πώς πισίλ. Ένα λεπτό. Τι έκανα. Πώς πισίλ. Είπα λάθος το όνομά σας. Κυρία Πρόεδρε, ακολουθώ και υποστηρίζω την πρόταση. Υπάρχουν πολλά θετικά, όπως την ηλεκτρονική ψήφο. Θέλω όμως να κρούσω κόδωνα κινδύνου να, για την ε, η ε, ενδυνάμωση ε, του ευρωπαϊκού, της ευρωπαϊκής διαργασίας των εκλογών. Πρέπει να παραμείνουν στο εθνικό πλαίσιο οι ευρωεκλογέ. διότι αν επιβάλλουμε κάποια θέματα, κάποιες, κάποιους και προϋποθέσεις, τότε θα διαρρήξουμε τη σύνδεση μεταξύ πολιτών και εκπροσώπων και θα πρέπει πραγματικά οι πολίτες να μπορούν και να γνωρίζουν ποιους εκλέγουν στο Ευρωκοινοβούλιο, να κατανοούν τη γλώσσα γλώσσα και να ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Αν διαρρήξουμε αυτό το σύστημα τότε πολλά αρνητικά θα υπάρξουν ως επιπτώσεις. Δεν θα γνωρίζουν καν ε, ε τους ε ε, ε, ε, βουλευτές τους οι μικρότεροι. Διαδικασίας επιχείρησε να κατασκευαστεί ο περίφημος Ευρωπαϊκός Δήμος, European Demos έτσι με την τροπολογία ένα καθορίζεται ότι τα μέλη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου εκλέγονται ως αντιπρόσωποι των πολιτών της ένωσης και όχι ως εκπρόσωποι των λαών των κρατών μελών της ένωσης. όμως οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν μπορούν να καταργηθούν με νόμους και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. επιπλέον με το νέο εκλογικό νόμο επιβάλλεται κατώτατο όριο τρία για την κατανομή των εδρών με στόχο να αποκλειστούν από την επόμενη σύνθεση της ευρωβουλής διάφορα κινήματα και ενοχλητικές φωνές κατά της γερμανικής ευρώπης για τον νέο εκλογικό νόμο επίσης ενισχύεται με αυτόν η ευρωπαϊκή κομματοκρατία σε βάρος των κινημάτων και των πολιτών. ταυτόχρονα υπονομεύονται οι λαοί ως πηγή δημοκρατικής νομιμοποίησης ενώ το παζλ του ευρωπαϊκού melting pot συμπληρώνει η παράγραφος 21 της έκθεσης που αμφισβητεί τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών της ένωσης και ζητά εκπροσώπηση μειωνοτικών γλωσσών στις ευρωπαϊκές εκλογές. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η νέα μεταρρύθμιση δεν πρόκειται να ενισχύσει τη δημοκρατική διάσταση ούτε την νομοθετική ε, την, μάλλον, ούτε θα νομιμοποιήσει τη δημοκρατική εκλογή ούτε θα βοηθήσει στην ε, ηθαγένεια ε, δίνει μόνο βοήθεια σε κόμματα ή συνασπισμούς μιας, ενός έθνους και ενός αλλά όχι στις περιφερειές. Πρόκειται για κάτι το υποχρεωτικό που είναι κατά των μειονοτήτων και θέλει να εξορίσει ε, τους εκατομμύρια πολίτες από το πολιτικό παιχνίδι της Ευρώπης. Καθόλου πιο δημοκρατικό ούτε πιο αποτελεσματικό όπως ε, ισχυρίστηκαν οι, οι, ε, Αν θέλουμε περισσότερη νομιμότητα στη χώρα μου και στην Ευρώπη θα έπρεπε να μπορεί κανείς να εκλεγεί με μία μοναδική περιφέρεια περιφέρεια, από μία μοναδική περιφέρεια. Η ε, κυρία Ρίγα, ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω πως αυτή η πρόταση ε, είναι σίγουρα μια χαμένη ευκαιρία Εάν δούμε την, την τρέχουσα κατάσταση, όλοι οι Γερμανοί ευρωβουλευτές θα ήταν πρόθυμοι να στηρίξουν οποιαδήποτε πρόταση για εκλογική νομοθεσία για να μπορέσουν να πιέσουν για αυτό το κατόφλι. Χρησιμοποιήστε λοιπόν αυτήν την δυνατότητα για μια φιλόδοξη πρόταση που θα συμπεριλαμβάνει διακρατικές, διακρατικά ψηφοδέλτια. Πρέπει να βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση, αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνουμε μόνο χρόνο βάζοντας το λογότυπο του Ευρωπαϊκού Κόμματος ή αποκλείοντας τα μικρά κόμματα από το Ευρωκοινοβούλιο. Θα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι ευρωβουλευτές από τις διάφορες χώρες θα ενθαρρυνθούν να συνεργαστούν μέσω κοινών πολιτικών θέσεων που θα προτάξουν. Αυτό θα μπορούσαμε να το πετύχουμε με διακρατικά ψηφοδέλτια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φιλοδοξία σε αυτή την πρόταση. Είναι μια προσπάθεια για να εξαλειφθούν τα μικρά γερμανικά κόμματα από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Qui Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι εξεπλάγει όταν άκουσα κάποια από τα σημερινά σχόλια. Το κατώτατο αυτό όριο αναφέρθηκε επανειλημμένα το γερμανικό συνταγματικό δικαστηρίο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ελάχιστο κατόφλιο ήταν κάτι απαράδεκτο. Σέβομαι την αποφασή του, όμως μπορώ να σας πω ότι συνταγματικό δικαστήριο στην Τσεχική Δημοκρατία και αυτό κατέληξε σε μια απόφαση από αυτού και αποφάσισε να διατηρηθεί το κατώτατο όριο διότι δεν θεωρήθηκε κάτι αντισυνταγματικό. Έχουμε δύο διαφορετικά συνταγματικά δικαστήρια να αποφασίζουν ποικιλοτρόπω προ αντίθετε κατευθύνσει. Βλέπετε τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να το καταλαβαίνετε. Τα, τα συνταγματικά δίκαια των διαφόρων κρατών ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχουν διαφορετικούς κανόνες. Και νομίζω ότι αυτού του είδους οι διαιρέσεις δεν είναι κάτι καλό. Λοιπόν, θα ήμουν πάρα πολύ προσεκτική ε, όσον αφορά τη θέσπιση των κοινών κανόνων. Πρόεδρε, είναι σαφές ότι είναι αντιδημοκρατική φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δούμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Αποφεύγονται τα δημοψηφίσματα ή δεν γίνονται σεβαστά τα αποτελέσματά τους όταν δεν είναι βολικά. Ε, όταν κανένας δεν μπορεί να εγκρίνει τις συνθήκες, ε, αλλάζουν οι ίδιες, ε, ισχύουν οι κανόνες χωρίς να εγκριθούν καν αυτές οι συνθήκες. Αυτό που είπε η ίδια η κυρία κυρια Μέρκελ ε, δικαιολογώντας ε, ε, αιτιολογώντας τις αποφάσεις τους. Καθορίζονται οι κυβερνήσεις, επιβάλλονται πολιτικές ε, τα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα ε, υποτάσσονται όπως η, τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν υπάρχει δυνατότητα να το κρύψουμε πια. Είναι αντιδημοκρατική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα ε, οικοδόμημα που είναι διαρθωτικά αντιδημοκρατικό. Σε αυτήν εδώ την έκθεση περιλαμβάνονται πολύ σημαντικά και σοβαρά προβλήματα. Πρόκειται για ακόμα μια αντιδημοκρατική κλιμάκωση. Ε, τελείωσε ο χρόνος σας, λυπάμαι, ε, διακόπτη η Πρόεδρος. Κυρία Κρέτσου, στρέφομαι και πάλι σε εσά αφού τελείωσε το κατδιάι. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας και για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ θέλω να κλείσω επαναλαμβάνοντας ότι η Κομισιόν στηρίζει πλήρως στις προσπάθειες του Κοινοβουλίου για την υιοθέτηση αυτής της επίκαιρης και φιλόδοξης έκθεσης. Κατά τη γνώμη μας, έτσι θα υπάρχει μια ένωση, μάλλον για να υπάρχει μια ένωση δημοκρατικών αλλαγών θα πρέπει να βελτιώσουμε τη δυνατότητα της, τη διαδικασία εκλογής των υποψηφίων. Θέλουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό δημοκρατικό σύστημα όπου οι πολίτες θα συμμετέχουν πλήρως. Η ενίσχυση της σχέσης ανάμεσα στις εκλογές των εκπροσώπων των πολιτών και την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για, την, για, για το εκτελεστικό όργανο mm. της ε, Ένωσης ε, σημαίνει ε, συμμετοχή και των πολιτών, όπως το είπα και στην αρχή. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε τις ποσοστώσεις και την ισορροπία του φύλου, των φύλων, πράγμα το οποίο εσείς υποστήριξα ως Ευρωβουλευτής. Η πρόταση αυτή νομίζω πως είναι ένας ε, συγκεκριμένος τρόπος για να δημιουργηθεί νέο είδος ενδέσμευσης και συμμετοχής στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και να κινητοποιηθούν έτσι οι πολίτες να παίξουν πιο δραστήριο ρόλο στην ευρωπαϊκή δημοκρατία. Όπως είπα εξ αρχής, αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμο να οικοδομήσουμε και να συμβάλλουμε στην εμπιστοσύνη των πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ. Επανερχόμαστε στους ε, εισηγητές. Η κυρία Χιούμπνερ, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους είπαν ότι μας λείπει η φιλοδοξία, αλλά και όσους ε, λένε ότι είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι. Φυσικά αυτές οι ομάδες είναι σε αυτή την αίθουσα. Για όσου λένε ότι δεν ήμασταν αρκετά φιλόδοξοι με την έκθεση αυτή, θα ήθελα να πω ότι κάποιε φορέ στην εργασία μα και όλοι το είναι, έχουμε αυτή την εμπειρία, θέλουμε να έχουμε περισσότερο κόσμο να συμφωνεί με τις ιδέες μας, που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικέ για του Ευρω... για και μετά η φιλοδοξία μα έρχεται στο κοινό επίπεδο φιλοδοξία όλων και αυτό σε κάποιο βαθμό εξηγεί γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Δεν μπορούσαμε επίση να τα επιτύχουμε γιατί υπάρχουν και διαδικασίε με το Συμβούλιο δεν Πρέπει να ε, πάει αυτή η πρόταση στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο θα αγνοήσει τελείως ε, μπορεί να αγνοήσει τελείω την πρότασή μα. Γι' αυτό και προσπαθούμε να βάλουμε κάτι που θα περνούσε από όλο το σύστημα και που θα μπορούσε να μα πάει να βήμα μπροστά στην εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο δικαίωμά του να αποφασίζει για την εκλογική του την διαδικασία. Σε κάποιο βαθμό λοιπόν ίσως αυτό να εξηγεί το πρώτο, την πρώτη ομάδα σχολείων. Αλλά για όλους όσους λένε ότι προχωράμε υπερβολικά πολύ, να πω ότι διαφωνώ απολύτως μαζί σας και όταν λέτε ότι έχουμε προχωρήσει πολύ γιατί έχουμε αναλάβει ευθύνη για θέματα που θα έπρεπε να μείνουν στο εθνικό επίπεδο και στην εθνική κυριαρχία, σε αυτό το επίπεδο της διαδικασίας, θα ήθελα να πω ότι η πρόταση αυτή φέρνεται ως ευρωβουλευτές πιο κοντά στους ψηφοφόρους τους. Έρχονται οι Ευρωπαίοι πολίτες πιο κοντά στην Ευρώπη και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αδυναμία της Ένωσης ε, ε, μεγάλη απόσταση, τεράστια απόσταση ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες και την Ένωση. Ε, ελπίζω λοιπόν ότι μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε στο επίπεδο της Επιτροπής εδώ και θα συνεχίσουμε και με το Συμβούλιο να συζητάμε ότι ως αποτέλεσμα θα έχουμε κάτι που ίσως να μην είναι και μεγάλο ορόσημο όπως λέγει η Επίτροπος αλλά πάντως θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε μπροστά σε αυτό το μονοπάτι για ε, τον καθορισμό της εκλογικής διαδικασίας ε, μας εδώ στο Κοινοβουλίο. Όπως έλεγε ο κύριος Σέφλιν, είμαστε μάλλον το μοναδικό κοινοβούλιο στον κόσμο που δεν μπορεί το ίδιο να αποφασίσει για την εκλογική του διαδικασία. Τέλος, για το κατόφλι και το γερμανικό ε, συνταγματικό δικαστήριο, ελπίζω πως ο Γιολάινα θα το εξηγήσει, αλλά από ό,τι θυμάμαι το συνταγματικό δικαστήριο είπε επίση ότι εάν υπήρχε ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κατόφλι, τότε θα ήταν διαφορετική υπόθεση. Και γι' αυτό και προτείνουμε ευρωπαϊκό κατόφλι, για να αποφύγουμε όλα τα προβλήματα που έχουμε σε εθνικό επίπεδο με τις διαφορετικές ερμηνείες των διαφόρων συνταγματικών δικαστηρίων. Πάντως ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι και ελπίζω ότι θα έχετε το χρόνο να σκεφτείτε πώς θα ψηφίσετε. Λάινεν ο εισηγητής. Ο κύριος Λάινεν, μάλιστα και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ όσου συμμετείχαν στη συζήτηση. Ο συνάδελφο Σέπφλιν πράγματι είπε ότι ένα ελάχιστο κατόφλι βαίνει καλός, αλλά να μην είναι υπερβολικά υψηλό. Ε, αυτό κάναμε. Είδαμε τι συμβαίνει στα 26 κράτη-μέλη <clears throat> παντού νομοθετικά ή de facto υπάρχει ελάχιστο κατόφλι 3%. Και τώρα για δύο επιπλέον κράτη όπου δεν υπάρχει τέτοιο κατόφλι προτείναμε να ισχύει αυτό. Αυτό είναι ο κανόνας στις περισσότερες από τις χώρες μας και έχει, είναι συν, συνήθις αυτός ο κανόνας, έχουν εξοικειωθεί με αυτόν οι πολίτες και έτσι λειτουργεί σωστά. Και πράγματι συνάδελφοι, το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο στην ομολογία του αυτή την απόφαση έλαβε. Άνοιξε όμως το κατόφλι, την πόρτα για ένα ελάχιστο κατόφλι. Είπε, εφόσον δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ευρωπαϊκό εκλογικό δίκαιο σχετικά με αυτό, το κάνουμε αυτό, το θεσπίζουμε για τη χώρα μας. Και πρέπει να παρακολουθηθεί η εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις νέες αρμοδιότητες του για την εκλογή του εκτελεστικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο επιτελούμε με την εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τότε θα άλλαζε και η προσέγγιση με το μηδενικό κατόφλι. Αυτά είναι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η άλλη πλευρά. Το κατανοώ για τα πολύ μικρά κόμματα, αλλά δεν είναι σωστό να υπάρχει τέτοια μονομερής παρουσίαση των πραγμάτων με τέτοια επιχειρήματα. Με ενθαρρύνουν συνάδελφοι που είπαν ότι θα έπρεπε να είχαμε πάει λέει, πολύ πιο μακριά. Θεωρήσαμε όμως με βάση την πείρα από την τελευταία περίοδο ότι θα πρέπει σε δύο βαθμίδες, σε δύο κλίμακες να κινηθούμε. Η πρώτη βαθμίδα, η κλίμακα τώρα, σήμερα, εφόσον είναι εφικτό. Και στη συνέχεια θα υποβάλουμε περαιτέρω προτάσεις σε μια περαιτέρω βαθμίδα μέσω μιας μεγαλύτερης, σε μια μεγαλύτερη διαβούλευση με τις ε, κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών για να προχωρήσουμε παραπέρα. Ας μην αυταπατώμαστε. Ευρωπαϊκοί ε, εκλογικοί συνδυασμοί και λίστες ε, απαιτούν τροποποιήσεις ε, σε σχέση με τα πράγματα όσα έχουν σήμερα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σήμερα, το έδειξε η πείρα από την πρώτη προηγούμενη περίοδο. Είναι ένα ορόσημο αυτό, όπως ανέφερε η κυρία Επίτροπος Κρέτσου, σε σχέση με τις δεκαετίες που δεν έγινε τίποτα κατά το παρελθόν. Είναι ένα μεγάλο βήμα μάλιστα προς τα εμπρός και δεν θα έπρεπε να δηλιάσουμε να το κάνουμε. Πώς να το πω, δεν πρέπει να απολέσουμε την ευκαιρία <clears throat> διότι αν απολέσουμε την ευκαιρία δεν θα υπάρξει μεταρρύθμιση του εκλογικού πλαισίου και το 2019 πάλι με τον παλαιό τυφλοσούρτη θα προχωρήσουμε που είναι ελληματικός ούτως ή άλλως. Τελευταία παρατήρηση. Εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται, ναι μεν στις χώρες μας, στα κράτη-μέλη να γίνονται εκλογές, αλλά εδώ όταν βρισκόμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο να εκπροσωπούμε το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όλα και όχι τα κράτη-μέλη μας, ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ευρωσκεπτικιστές στην Ευρώπη και μπορούμε να κάνουμε όποιες προτάσεις θέλουμε, αλλά ε, εις ε, ότα κοφών. Και είναι μια μειονότητα και θα παραμείνουν μειονότητα αυτοί οι ευρωσκεπτικοί σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει